Κύριε Πόσελ, θέλετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σας εκτιμώ πάρα πολύ και η Προεδρία σας ήταν πάρα πολύ καλή σε αυτή την ψηφοφορία. Μόνο μία παράκληση έχω προς όλους τους αντιπροέδρους την Πέμπτη το μεσημέρι να μην εύχεστε καλό Σαββατοκύριακο σας παρακαλώ. Έχουμε και το απόγευμα κατεπήγοντα, έχουμε ψηφοφορίες, είναι πλήρε και έγκυρες ακόμα και αν πολλοί ταξιδεύουν. Σας παρακαλώ μην ε, λέτε τέτοια πράγματα πριν το τέλος της συνόδου που είναι στις 5 ώρα το απόγευμα και μην εύχεστε καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο τώρα, γιατί είναι η τελευταία ευκαιρία για εμένα να το πω. Δεν εννοώ ότι τελειώσαμε. για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι σε αρκετές χώρες το έργο της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γίνεται δυσκολότερο εξαιτίας των νομοθετικών ή διοικητικών κανόνων και ορισμένες φορές γίνεται ακόμη και αδύνατο εξαιτίας φυλακίσεων και άλλων απειλών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που πάντα υπεραμείνεται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίω, νομίζω ότι θα έπρεπε μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρμοδιοτήτων που της δίνει η νέα συνθήκη της Λισαβόνας να προσφέρει μεγαλύτερη ευρωπαϊκή καθοδήγηση και συμπερίληψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις διμερείς συμφωνίες εμπορικές και άλλες με τρίτες χώρες. Ακόμη και για την αξιολόγηση των τρίτων χωρών προκειμένου να υπάρξουν εμπορικές συμφωνίες αλλά και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η έκθεση της κυρίας Χάουταλα είναι πολύ καλή και την ευχαριστώ. Αν όμως τα συμπεράσματα της έκθεσης ε, εφαρμοστούν, τότε η υπεράσπιση των ε, υπερμάχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βελτιωθεί πολύ και γι' αυτό υπερψήφισα την έκθεση. Μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι όλους τις υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να μην χρειάζεται να πεθαίνουν στο όνομα αυτών. Βίρ, για ένα λεπτό. Δεν είναι εδώ Ο κύριος Μπάτεν για ένα λεπτό. και ο κύριος Μπάτεν έχει φύγει. Έκθεση Κοέλιο. Ο κύριος Μαστέλλα, για ένα λεπτό. Ούτε ο κύριος Μαστέλλα είναι εδώ. Έκθεση Ρωμέβα Ιρουέδα, διάσταση του φύλου στο πλαίσιο οικονομικής ύφεσης. Πάλι η κυρία Οβίρ, αλλά δεν είναι εδώ. Είναι εδώ η κυρία Οβίρ, έχει επιστρέψει. Όχι. Η κυρία Οβίρ επίσης, στην έκθεση Φουγερέδο, Είναι εδώ η κυρία Οβίρ. Όχι. Ο κύριος Στάκουλα, στην έκθεση για τον αθλητισμό, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την έκθεση αυτή και την εισηγήτρια την κυρία Τόρι Πακ που είναι πρόεδρος της Επιτροπής μας. Είναι πολύ καλή η έκθεση, την υπερψήφισα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν κανόνες ηθικής και δεοντολογίας και στον αθλητισμό που πρέπει να επιβάλλονται, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ανύπαρκτη. Και από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι το εμπόριο ανθρωπίνων όντων, ποδοσφαιριστών. Και σε πολλές περιπτώσεις έχουμε ενδείξεις ε, ότι οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι καταχρώνται τις δυνατότητες αυτής. Θα πρέπει ο εθνισμός να είναι όσο γίνεται πιο καθαρός. Υποστήριξα λοιπόν την έκθεση της κυρίας Πακ και ελπίζω να κάνουμε κανόνες με τη FIFA και την UEFA. Ευχαριστώ. Στην έκθεση για τη συνάντηση κορυφής της Ευρώπης Ρωσίας, ο κύριος Πρέντα για ένα λεπτό. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ψήφισα διαφορετικά από την ομάδα μου για τις τροπολογίες 1 και 2 των πρασίνων στο κοινό ψήφισμα. Στήριξα αυτές τις τροπολογίες γιατί είναι πολύ σημαντικές ε, κατά τη γνώμη μου. Όταν αναλύουμε ε, τα αποτελέσματα του Συμβουλίου να δούμε την ε, γενικότερη κατάσταση στη Ρωσία και αυτό που προέκυψε είναι ότι οι υπέρμαχοι της ελευθερίας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στη Ρωσία. Η Ρωσία λοιπόν θα έπρεπε να αμήνεται του δικαιώματος για ισονομία και για δίκαια δίκη. Ο κύριος Κέλλαμ για ένα λεπτό. Thank you Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και η δική μου άποψη είναι παρόμοια. Στις τροπολογίες 1 και 4, 1 έως 4 για τη Ρωσία ψήφισα διαφορετικά. Είπαν κάποιοι ότι η επιχειρηματική σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας δεν θα έπρεπε να ασχοληθεί με όλα τα προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμως αυτά τα πράγματα συνδέονται. Και αν σκεφτείτε ότι υπήρξαν 40 διαδηλώσεις σε 40 ρωσικές πόλεις στις 31 Μαΐου πριν την αρχή της Συνόδου, ζητώντας το δικαίωμα του να και υπενθυμίζοντας και την, το θάνατο του Σεργέη Σανίσκη αλλά και την τροπολογία 3 που ζητάει να μην υπάρξει ασυλία για τους θανάτους ε, των υπερμάχων των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για όλους αυτούς τους λόγους ψήφισα διαφορετικά. Ο κύριος Προτασίεβιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Χάουτελα και τους συναδέλφους από τους Πρασίνους που κατέθεσαν τροπολογίας για την κατάσταση των υπερμάχων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Παρόλο που αυτό το θέμα δεν ήταν θέμα της Συνόδου, ψήφισα την τροπολογία 3 της κυρίας Χάουταλα γιατί θέλω ένα ψήφισμα που θα αντικατοπτρίζει τις απόψεις μας για την κατάσταση της Ρωσίας και τη σχέση της με τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. θέματα όπως τα θεμελιώδη δικαιώματα ή το δικαίωμα του συνέρχεστε θα έπρεπε να παραμείνουν σημαντικά στις σχέσεις μας με τη Ρωσία. και τον αποκλεισμό της Γάζας ο κύριος Χίγκινς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ απέσχον στην ψηφοφορία διότι το ψήφισμα δεν καταδικάζει αρκετά ε, τη βία που έχει εξαπολύσει και την επίθεση βίας που έχει εξαπολύσει το Ισραήλ κατά του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Εννέα ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων δολοφονήθηκαν. Και αυτό έχει αποτροπιάσει και αειδιάσει τον κόσμο ολόκληρο. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι το Ισραήλ ε, απορρίπτει την ανεξάρτητη έρευνα και ανάκριση. Και επίσης θα πρέπει να καταδικάσουμε και την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τον πρόεδρο Ομπάμα που δεν επέκρινε ε, την κατάσταση αυτή. Δεν μπορούμε να έχουμε καμία εμπιστοσύνη στον ΟΗΕ για ψηφίσματα για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Παντού έχουμε επιθέσεις και στο Τελαβίβ μεγάλη πορεία Παλαιστινίων και Ισραηλινών και οι εργαζόμενοι, η εργατική τάξη θα δώσει τη λύση εκεί στα προβλήματα στη Μέση Ανατολή. Σε μια δημοκρατική κοινωνία. Ευχαριστώ. για ένα λεπτό. Πρόεδρε, εγώ υπερψήφισα το ψήφισμα για την κατάσταση στη Γάζα, αλλά δεν με ικανοποιεί πλήρω η διατύπωση. Και βέβαια είναι σημαντικό να ακούγεται και η φωνή του Κοινοβουλίου για τα όσα συνέβησαν στι 31 Μαου. Βεβαίω και θα πρέπει να έχουμε αξιόπιστη διεθνή παρουσία και έρευνα θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δείξει το ενδιαφέρον του για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, αλλά υπάρχει και το θέμα της ασφάλειας του Ισραήλ και όλα αυτά ε, είναι ε, θέματα που αφορούν αυτά που λέει παράγραφος 2 για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου ή για συλλογικές τιμωρίες. Δεν, δεν μου αρέσουν αυτά που αναφέρει το ψήφισμα. Θέλουμε να παίξουμε ρόλο στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να είμαστε ουδέτεροι, διαμεσολαβητές και ανεπηρέαστοι. Δεν βοηθάει το ψήφισμα για την ειρήνη. Thank you again, President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στήριξα το ψήφισμα για τη Γάζα. Θεωρώ όμως ότι συναισθηματικά δεν είναι ιδιαίτερα ισορροπημένο. Ζητάμε αμερόληπτη διεθνή έρευνα του θέματος, αλλά δεν θα έπρεπε το μεταξύ να βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Και γι' αυτό ήμουν κατά του δεύτερου τμήματος, της παραγράφου 2 δηλαδή, που δηλώνει ότι επρόκειτο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Αυτό θα πρέπει να το διαπιστώσουν οι ερευνητές. Και επίσης ήμουν κατά της αιτιολογικής σκέψης γάμα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον κύριο Κέλλαμ. Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος όπως και η ομάδα μου, αλλά θέλω να πω ότι στο δικό μας ψήφισμα υπήρχαν σημαντικά σημεία που δεν αναφέρθηκαν. Για παράδειγμα, το ΕΛΚ ήθελε να αναγνωρίσει το δικαίωμα του Ισραήλ να έχει ασφαλή σύνορα. Αυτό είναι προφανές, αλλά δεν αναφέρθηκε στο τελικό ψήφισμα. Γιατί? Κύριο για ένα λεπτό. Ψήφισα κατά του ψηφίσματος, γιατί κατά τη γνώμη μου, δεν ήταν ισορροπημένο το ψήφισμα. Ήταν κατά του Ισραήλ και δεν κοίταζε την συνολική εικόνα. Κατά τη γνώμη μου η Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε εδώ. Θα έπρεπε να είχαμε αποφύγει την παρουσία πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον στολίσκο, γιατί στόχος του ήταν η πρόκληση. Υπάρχει διεθνές ναυτικό θαλάσσιο εμπάργκο σε αυτή την περιοχή. Γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτό από άποψη διεθνούς δικαίου. Εγώ από την τηλεόραση κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ο στόχος του στολίσκου ήταν να αντιπαρατεθεί στο Ισραήλ. Δεν μπορούμε να στηρίζουμε τέτοιες δραστηριότητες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Πρέπει να υπερασπιζόμαστε τα ανθρωπίνα δικαιώματα και το δημοκρατικό κράτος του Ισραήλ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στο ψήφισμα αυτό εκφράζεται θεμητή κριτική ε, στη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ. Δυστυχώς όμως μένουμε μόνο στα λόγια, δεν περνάμε στα έργα. Αν ήταν οι Κουβανοί ή οι Ιρανοί που είχαν επιτεθεί σε διεθνή ύδατα, σε ευρωπαϊκά σκάφη και είχαν σκοτώσει ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φανταστείτε τι θα είχε γίνει τότε. Αυτό τι σημαίνει. Θα έλεγαν ότι είναι τρομοκρατία αυτό το πράγμα. εδώ έχουμε καθεστώς προνομιακών εμπορικών σχέσεων με το κράτος αυτό. Δεν μπορεί να διατηρηθεί. Δεν θα το κάνατε και με τις άλλες χώρες αν γινόταν αυτό. Θα είχαμε τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Το πρόβλημα με το ψήφισμα είναι ότι τα λέει ωραία ε, και ε, συμπαθητικά, αλλά δεν οδηγεί σε καμία δράση. Και η προνομιούχα σχέση με το Ισραήλ επίσης δεν διαρριγνύεται. Αν θέλει το Κοινοβούλιο να παραμείνει αξιόπιστο, θα πρέπει να δράσουμε κιόλα. Ευχαριστώ. Η κυρία δεν συμμετείχα στη ψηφοφορία γιατί το κείμενο περιείχε τόσα λάθη επί της ουσίας που δεν θα έπρεπε καν να υφίσταται. Οπότε συμφώνησα με το ΕΛΚ και τον κύριο Τάκουλα που λένε ότι η καταδίκη του Ισραήλ και αναφορά ότι παραβίασε το διεθνές δίκαιο χωρίς να έχουμε τα αποτελέσματα της έρευνας την ίδια στιγμή που ζητάμε να υπάρξει αμερόληπτη διεθνής έρευνα είναι κάτι το οποίο ήταν λανθασμένο και μη ρεαλιστικό. Επίσης χρησιμοποιούμε διαφορετική γλώσσα για τους πολίτες και τις αρχές του Ισραήλ από ό,τι για τους ακτιβιστές. Κάτι που δημιουργεί αδικαιολόγητη φόρτιση. Ο κύριος Βιγγένιν για δύο λεπτά. Δεν είναι παρόν ο κύριος Στην έκθεση για τις πλημμύρες στις χώρες Κεντρικής Ευρώπης, ο κύριος ε, Μεστσάρος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα στη κεντρική και ανατολική Ευρώπη η κατάσταση είναι ολέθρια, καταστροφική, μετά από πλημμύρες. Έχουν υπερχειλήσει τα ποτάμια ε, και χρειαζόμαστε επιγόντως βοήθεια. Πολλοί κόσμος έχει χάσει το βιώσει το ολόκληρο. Χαίρομαι πάρα πολύ που αναγνώρισε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Γι' αυτό θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να υπερψηφίσουμε και το γεγονός ότι υπερψηφίσαμε αυτό το ψήφισμα. Θα ήθελα να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα να βοηθήσει επιγόντως οικονομικά τους πολίτες Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Αγαπητοί συνάδελφοι, η συνεδρίαση διακόπτεται ως ώρα.